Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Αύριο στι 9 ξαναρχίζουμε. Είναι διαθέσιμη η ημερήσια διάταξη στο site του Κοινοβουλίου. Καλό σα βράδυ, καλή σα νύχτα.